με συγκεκριμένες προτάσεις όταν συγκεκριμενοποιηθούν τα νομοθετικά κείμενα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και με την παρέμβασή σας ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση και επανερχόμαστε στην ε, ημερήσια διάταξη. Τώρα έχουμε μια άλλη ε, προφορική, ε, προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τις εμπορικές συμφωνίες κατά των απομιμήσεων. Κύριε Ντεχούχτε, καλώς ήρθατε και θα δώσω το λόγο στο συντάκτε στους προφορική της ερώτησης που είναι έξι. Καταρχάς ο κύριος Σλίτερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να υπερασπίσουν το ρόλο τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και ε, να ε, υπάρξει εφαρμογή των συμπεφωνημένων και εδώ πρέπει να διαφυλάξουμε και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Διαφορετικά αυτό το θεσμικό όργανο δεν μπορεί ούτε να παίξει το ρόλο που πρέπει, ούτε να ανταποκριθεί στις προσμονές των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει πρόσβαση εις ε, τα ε, έγγραφα και ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί το λόγο της. Πολλοί πολίτες ανησυχούν για την ελευθερία της εκφράσεως διότι υπάρχουν πολλές νομοθεσίες οι οποίες περιορίζουν τις ελευθερίες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρχει σεβασμός των Πού είναι η διαφάνεια. Ίσως το περιεχόμενο είναι ε, λίγο ευαίσθητο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας πει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξει διαφάνεια και ε, για να μπορέσουμε να υπεραμεινθούμε των ε, δικαιωμάτων μας. Μόνο όταν όλα αυτά είναι ξεκαθαρισμένα θα μπορέσουμε να προβούμε σε διαμόρφωση διατάξεων, σε σύναψη συμφωνιών, διότι τώρα υπάρχει μία παράδεκτη κατάσταση όπου και κλεισμένων των θυρών πρέπει να ρωτάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι υπάρχει σε μία συμφωνία. Οι, πολιτικοί, οι πολίτες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ψάχνουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές στα σύνορα και ότι θα μπορούν να κυκλοφορήσουν κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Πρέπει να δεσμευτείτε σήμερα ότι θα υπάρξει πλήρη ε, ελευθερία διότι διαφορετικά θα απαντήσω με την κλασική έκφραση ότι θα τα πούμε στα δικαστήρια. Κάσπαρη, δύο λεπτά. Ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ε, ε, ε, υπάρχουν θέματα πνευματικής ιδιωτικησίας αλλά και άλλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν μεγάλη σημασία βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραποιήσεις και βλέπουμε ότι φτάνουν σε ένα ύψος 250 δισεκατομμυρίων ευρώ αν πρόκειται δε για ε, ένα φάρμακο μπορεί να είναι πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις, δηλαδή ο άνθρωπος να μπορεί να πεθάνει από ένα παραποιημένο φάρμακο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, ταχθούμε κατά της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας διότι δεν είναι δυνατόν να κατάσχουμε στα σύνορά μας 850 εκατομμύρια παραποιημένα εμπορεύματα εκ των οποίων ορισμένα θέτουν σε κίνδυνο και την, και υγεία των πολιτών. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας εμπλεκόμαστε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν γι' αυτό θα θέλαμε στις επόμενες εβδομάδες και μήνες μεγαλύτερη διαφάνεια να ξέρουμε ακριβώς ε, τι ε, ε, γίνεται με τις διαπραγματεύσεις να ε, συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να υπάρξει μια συνεκτική συμφωνία αλλά προς συμφέρον των εργαζομένων, των εργοδοτών, των βιομηχανιών να υπάρξει μια σωστή συμφωνία η οποία όμως συγχρόνως σας και το κοινωτικό εκτιμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κασπάρη. Λάγκε, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ, με μένα με απασχολούν τρία ερωτήματα. Το ένα από αυτά είναι ε, γιατί δεν υπάρχει ακόμη διαφάνεια εφόσον από 1η Δεκεμβρίου ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και ε, το Φεβρουάριο συνάψαμε μία διαθεσμική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Συμβούλιο είναι παρατηρητής και το Κοινοβούλιο δεν ε, εμπλέκεται και τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα δημόσια. Δεύτερη ερώτηση. Ε, ποιος διαπραγματεύεται για τη συμφωνία αυτή άκτα, δηλαδή για την καταπολέμηση της παραποίησης. Δεν είναι ε, όπως τα τρίψ εις τον ΠΟΕ, αλλά εδώ πρόκειται για μεμονωμένα κράτη και ακούμε ότι υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών και σημαντικές βιομηχανίες. Δεν πρέπει να υπάρχουν τα ίδια μέτρα και σταθμά για όλους οι οποίοι κάθονται γύρω από το τραπέζι και διαπραγματεύονται. Και το τρίτο ερώτημα κύριε Πρόεδρε είναι ουσιαστικά γιατί διαπραγματευόμαστε, ποιο είναι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει σεβαστό το κοινοτικό και κτημένο. Εάν όμως δω τα έγγραφα που κυκλοφορούν έχω αμφιβολίες διότι μπορώ να καταλάβω ότι στις διαπραγματεύσεις μπορούν να υπάρξουν φραγές εις το διαδίκτυο προς το κοινό συμφέρον ότι μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί για την έρευνα και την επιστήμη μπορώ να καταλάβω ακόμη και ότι ορισμένοι θέλουν να εφαρμόσουν γενικευμένα συστήματα επιτήρησης. Αλλά πού είναι το κοινοτικό κεκτημένο σε όλα αυτά. Δηλαδή το lost profit, το χαμένο ο κέρδος πρέπει επίσης να τύχει της διαπραγματεύσεως ε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι αντάξιο των πολιτικών μας πεπιθήσεων και τέλος τι γίνεται με το online και offline. Δηλαδή διαβάζω ότι και το online και το offline αποτελούν μέρος του ψηφιακού κόσμου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει κανείς να ψάχνει τα λάπτοπ όταν ε, διέρχεται κάποιος στα σύνορα. Θα ήθελα απαντήσεις σε αυτές αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Νικόλα Ρινάλδη, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε συνάδελφοι. Είναι κρίμα ε, που συζητάμε αυτό το θέμα με... και είναι κρίμα που διαπραγματευτήκαμε με μυστικότητα μέχρι στιγμής. Υπάρχει ασυμμετρία. Η αμερικανική ε, βιομηχανία είχε πρόσβαση σε διάφορες ε, πληροφορίες διαφορετικά ήταν τα πράγματα όμως στην Ευρώπη ε, και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται, το έχουμε ξανασυναντήσει και αλλού. Ε, Παραδείγματο χάρη μιλήσαμε για τη συμφωνία με την Κορέα. Και τώρα αυτή η ιστορία με την εφαρμογή της συνθήκης ε, της Λισαβόνας θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η έλλειψη διαφάνειας. Ε, και νομίζω ότι αυτό το κρίμα ε, μας οδηγεί Μα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Ούτως ή άλλως αυτή η μάχη που δίνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ιερή. Εγώ προέρχομαι από μια ε, πόλη που τη γνωρίζετε ε, πολύ καλά κύριε Επίτροπε, ε, τη Βενετία. σκεφτείτε τα κρίσταλα Μουράνο ε, εμείς φτάναμε στο παρελθόν μέχρι και στη θανατική ποινή για όσους απομιμούνταν αυτά τα κρίσταλα. Ε, σε μια όλο και πιο παγκόσμια οικονομία αυτά τα εγκλήματα είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές απειλές. Ε, αυτή η συμφωνία δημιουργεί τεράστια προβλήματα και ε, χτυπάει καμπανάκια στην κοινή γνώμη και νομίζω τα ξέρει όλα αυτά τα πράγματα η Κομισιόν. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Αλλά νομίζω ότι και η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών θα πρέπει να ασχοληθεί. Μας απασχολούν τα θέματα, μας απασχολεί η ελευθερία ενημέρωσης ε, και πληροφόρησης μέσω του ίντερνετ, ε, το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα, ε, κάποιες, κάποια θέματα και κάποιες επιπτώσεις για τους service provider, ε, θέματα αστικού και ποινικού δικαίου, επομένω προσοχή Κομισιόν. Σα καλώ να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο να με διαβεβαιώσει μάλλον μήπως αν το άκτα θα χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσουμε, ε, για να παρεμποδίσουμε μάλλον την πώληση α, γενώσιμων φαρμάκων που δεν προστατεύονται από το copyright, αλλά που τα παράγουν ε, αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία και η Βραζιλία και μπορεί να ενοχλήσουν πάρα πολλές ε, μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Ευχαριστώ κύριε Ρινάλντι. Δυόμιση λεπτά ο Χέλμουντ Σόλτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πέτροπε Ντεγκόχτ. Όταν ε, συναντάστε ε, με τους εκπροσώπους μεγάλων κυβερνήσεων για να εφαρμόσετε ε, τις διατάξεις αυτών των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να εκπλήσεστε που δημιουργούνται ερωτήματα και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν τι διότι πρέπει και εσείς να καταλάβετε ότι ανησυχούν ε, οι διάφορες πολιτικές ομάδες για τα θέματα αυτά δηλαδή υπάρχει μία διαπραγματευσή όπου πρέπει κανείς να διασφαλίσει τα δικαιώματα του πολίτη, τη δημοκρατία της επικοινωνίας, την ε, αποκέντρωση, την, ε, τα θέματα των προσφυγών, προσωπικών δεδομένων τον του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό και θα σας παρακολουθούμε συνέχεια. Μια τέτοια συμφωνία θα έχει επιπτώσεις παγκόσμιες. Αλλά ε, η συζήτηση αυτή γίνεται χωρίς την εμπλοκή των υποανάπτυξη χωρών, της κοινωνίας των πολιτών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δηλαδή όλων των ε, ενδιαφερομένων που θα έπρεπε να σας θα πρέπει να προσπαθείτε να ε, βάλετε όλα τα αποτελέσματα μέσα σε δύο σελίδες και ε, δεν είναι δυνατόν ε, να προχωρήσετε έτσι. Πρέπει να μας αποκαλύψετε τα ίδια έγγραφα τα οποία δίνετε και στα κράτη-μέλη διότι εάν κάνουν ονειρεύεστε κάποια μέρα να ζητήσετε την συνέχεια λιμένες του Κοινοβουλίου θα πρέπει από πείρα να γνωρίζετε ότι πρέπει να, συμφω... να συμμορφωθείτε προς τις δημοκρατικές αρχές. Εάν δεν υπάρξει συζήτηση δεν πρόκειται να υπάρξει και απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Σαγιέτ Καμάλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω, Επίτροπε, μπορείτε να δείτε ότι πώ έχουν τα αισθήματα όλων των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Παρά τις ε, ιδεολογικές μας διαφορές και τις διαφορέ προσέγγιση που έχουμε σε αυτό το θέμα, όλοι συμφωνούμε για την ανάγκη μεγαλύτερη διαφάνεια. Νομίζω ότι και ελπίζω ότι αυτό το καταλάβατε. Όταν γίνονται διαπραγματεύσει και δεν επικρατεί επαρκή διαφάνεια, δεν καταλαβαίνουμε ποιε είναι οι αρχέ και ποια είναι η διαπραγματευτική μα θέση. Και Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δημιουργείται ένα κενό. Και οι φήμες γεμίζουν αυτό το κενό, οι διαρροές περί επισήμων εγγράφων. Δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι, αν, αν αυτές οι διαρροές εκφράζουν την πραγματικότητα ή όχι. Και βέβαια δεν μοιράζετε τις πληροφορίες σας μαζί μας. Και νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα σε ένα βαθμό. Δεν θέλουμε οι συνομιλητέ μα να ξέρουν το 100% τη θέση μα. Αυτό που ζητάμε όμω είναι μια λογική διαφάνεια. Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτέ τι πληροφορίε. Αν δεν θέλετε να μα δώσετε τα έγγραφα αυτά καθ' αυτά, δώστε μα κάποια σύνοψη. Εξηγήστε μα ποιε είναι οι αρχέ πάνω στι οποίε βασίζεται η διαπραγμάτευση. Για παράδειγμα, θα υποστηρίξουμε την πρόταση που από ό,τι φαίνεται συζητείτε, τα MP3 και τα laptops να μπορούν να κατασχεθούν στα σύνορα. Θα συμφωνήσουμε με την επιβολή κυρώσεων. Θέλουμε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η θέση μας. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν επί ενός κοινού κειμένου. Συνεπώς, το μπαλάκι είναι στη δική σας μεριά, να δείξετε διαφάνεια και να αναγνωρίσετε ότι μας χρωστάτε εξηγήσει και λογαριασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καμάλ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Κάραλντε Χούχτ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας για τις διαπραγματεύσεις άκτα. Να υπενθυμίσω καταρχήν ότι διαπραγματευόμαστε αυτή τη συμφωνία για να βελτιώσουμε την προστασία της καινοτομίας ε, το Made in Europe ε, τα, και όλους τους τομείς όπου μπορεί να παραβιαστούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστική καινοτομία θα πρέπει να έχουμε καινοτομίε, ε, είμαστε δημιουργικοί και να έχουμε και δικαιώματα αποκλειστικότητας. Είναι ένα από τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματά μας στην παγκόσμια φορά. Χρειαζόμαστε τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προστατεύεται στις εξαγωγικές μας αγορές. Προσπαθήσαμε να θέσουμε αυτό το θέμα στις ε, πολυμερείς, ε, στα πολυμερή φόρα, στο ΜΠΟΕ και στον, ε, στην Οργάνωση Προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αλλά οι προσπάθειές μας αυτές ε, μπλοκαρίστηκαν από άλλες χώρες. Παρά την προσπάθειά μας για πραγματική παγκόσμια λύση, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε συμμαχίες και η τελική συμφωνία ε, θα ισχύει για τις χώρες που την έχουν προσυπογράψει. Μακάρι ε, περισσότερες χώρες και κυρίως οι αναδυόμενες ε, οικονομίες και χώρες να προσχωρήσουν. Όπως είπα και στην ακρόασή μου όμως, αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι εμπιστευτικές. Αυτό δεν είναι ασύνηθες. Οι διαπραγματεύσεις ε, απαιτούν ένα ελάχιστο βαθμό εμπιστευτικότητας, ούτως ώστε τα μέρη να αισθάνονται άνεση για να κάνουν παραχωρήσεις και να ε, βυθομετρήσουν ένα τον άλλον πριν να ε, μπουν σε μια τελική συμφωνία. Συμφωνώ βεβαίω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται επαρκώ για τι εξελίξει των διαπραγματεύσεων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε δύο τομεί να ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο και να πείσουμε του εταίρου μα να συμφωνήσουν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την πληροφορία προ το Κοινοβούλιο, σα έχουμε δώσει τι διαπραγματευτικέ κατευθυντήρε γραμμέ ε, πλήρεις ε, εκθέσεις για τους γύρους των διαπραγματεύσεων και τα γενικά έγγραφα που προκύπτουν από τη Γενική Διεύθυνση ε, Εμπορίου. Το κάναμε αυτό σύμφωνα με τη Συμφωνία Πλαίσιου. Επίσης, η άκτα συζητήθηκε πολλές φορές στην ΙΝΤΑ, στην Επιτροπή δηλαδή Διεθνούς Εμπορίου, τα τελευταία τρία χρόνια. Θα ήθελα επίση να προσθέσω ότι η Κομισιόν έχει οργανώσει και δύο ε, συνεδριάσεις τον Ιούνιο 2008 και τον Απρίλιο του 2009 για τις διαπραγματεύσεις αυτέ άκτα, ανοιχτέ σε όλε τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, τα ΜΜΕ και του πολίτε. Επίση, μια άλλη δημόσια ακρόαση θα γίνει στι 22 Μαρτίου στι Βρυξέλλε, του 2010 δηλαδή. Μπορεί να θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι επαρκέ, ε, ότι έτσι δεν σχηματίζεται μια πλήρη εικόνα για το που έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσει. Έχω ε, δώσει οδηγίε στι υπηρεσίε μου να σα ενημερώνουν, να ενημερώνουν όλου του βουλευτέ που ενδιαφέρονται για όλε τι πτυχέ των διαπραγματεύσεων. Επίση, ε, αυτέ οι πληροφορίε ε, θα υπάρχουν στη διάθεσή σα πριν και μετά από κάθε διαπραγματευτικό γύρο. Επίση, αναγνωρίζω ότι ο καλύτερο τρόπο για να ενημερωθείτε για τι συμβαίνει σε αυτέ τι διαπραγματεύσει είναι να διαβάσετε τα σχέδια διαπραγματευτικών κειμένων αυτό σα δίνει μια θαυμάσια εικόνα για το πού έχουμε φτάσει σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Όπω θα γνωρίζετε μάλλον υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των ε, μερών του ΑΚΤΑ ότι τα κείμενα αυτά τα διαπραγματευτικά δημοσιοποιούνται μόνο εφόσον συμφωνήσουν όλα τα συμβαλώμενα μέρη. Η Κομισιόν είναι υπέρ τη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων, το συντομότερο δυνατόν, όμω κάποιοι εταίροι μα στις διαπραγματεύσεις αντιτίθεται σε μια ε, δημοσιοποίηση πρόορη. Ε, διαφωνώ, αλλά δεν μπορώ μονομερός να σπάσω αυτόν τον κώδικα ε, ε, εμπιστευτικότητας. Γιατί πολλά διακυβεύονται. Πάντως, ε, σας διαβεβαιώνω ότι στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων τον Απρίλιο, η Κομισιόν θα πιέσει τους εταίρους να συμφωνήσουν στη δημοσιοποίηση των κειμένων για να και θα αντιμετωπίσουμε τα... και θα μιλήσουμε για τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου με τους εταίρους μας, κυρίως με τις ΗΠΑ. Είναι σημαντικό όλοι να γνωρίζουν τι διακυβεύεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, ακόμα πιο σημαντικό, να γνωρίζουν και τι δεν διακυβεύεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες σας για την ουσία, να υπενθυμίσω τις βασικές, τη βασική θέση της Κομισιόν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Καταρχάς, ο στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε ε, τις μεγάλες ε, παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων που έχουν σημαντικές εμπορικές επιπτώσεις δεν θα οδηγήσει σε περιορισμό των αστικών ελευθεριών ή σε προβλήματα για τους καταναλωτές. Δεύτερον, η άκτα αφορά μόνο την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν περιλαμβάνει τις ε, σημαντικές τροποποίησεις του δικαίου για την πνευματική ιδιοκτησία, παραδείγματο χάρη copyright ή τη διαδικασία, την ε, διάρκεια προστασίας ε, των δικαιωμάτων. Θα πρέπει να υπάρχουν όμως ελάχιστοι κανόνες για το πώς ε, εξασφαλίζουν τα, τα δικαιώματά τους στο δικαστήριο οι δικαιούχοι. το χάρη, οι Ευρωπαίοι σχεδιαστές όταν υπάρχουν ε, απομιμήσεις των δημιουργιών τους θα πρέπει ε, να είναι σε θέση ότι και στο εξωτερικό τα δικαιώματά τους θα εξασφαλίζονται και θα προστατεύονται. Επίσης, η άκτα θα πρέπει να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο ε, με το επίπεδο ε, εναρμόνισης ε, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες καθώς και το πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Δεν θα υπάρξει εναρμόνιση ή αλλαγέ στην κοινωτική νομοθεσία από, το, από την πίσω πόρτα ή το παραθυράκι. Με αυτή την έννοια η άκτα θα επηρεάσει τους Ευρωπαίους πολίτες γιατί δεν θα δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα χρειαστεί να, εφαρμο... να υπάρξει εφαρμοστική νομοθεσία. Όμως, ε, θα υπάρξει μεγαλύτερη προστασία για όσους καινοτομούν στις ξένες αγορές. Γνωρίζω τις ανησυχίες που εξέφρασαν κάποιοι από εσά για την εισαγωγή μιας υποχρεωτικής, του υποχρεωτικού κανόνα ε, των τριών χτυπημάτων ή της διαβαθμισμένης απάντησης ε, για την πειρατεία στο ίντερνετ κτλ. Θα πρέπει να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Ε, για να μην υπάρχει αμφισημία. Αυτός ο κανόνας των τριών χτυπημάτων είναι, δεν είναι υποχρεωτικό στην Ευρώπη. Οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την ευελιξία, ενώ παράλληλα θα σεβαζόμαστε τις αστικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υποστηρίξει την υποχρέωση μέσω της άκτα αποσύνδεσης λόγω παράνομου downloading. Επίσης, ε, δεν θα παρεμποδίζει άκτα την πρόσβαση στα γενώσιμα φάρμακα. Ξέρω ότι δημιουργούνται κάποια προβλήματα ε, για τις επιπτώσεις στα γενώσιμα. Ε, σας είπα και στην ακρόασή μου ότι όταν μεταρρυθμίσουμε τον, ε, την τελογενειακή νομοθεσία θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Επίσης ζητήσατε για μια ε, μελέτη αντικτύπου. Ούτως ώστε να μην ξεπεράσουμε το κοινοτικό κεκτημένο μέσω των, της άκτα. Θα βασιστούμε στις οδηγίες που έγιναν ε, το 2004 για την εφαρμογή του, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την πρόταση του 2005 για, την, εφαρμογή, για τις εφαρμοστικές διατάξεις για το IPR, τα δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Επίσης, ε, τη μελέτη του ΩΣΑ του 2008 για την απομίμηση και την πειρατεία. Αυτή η μελέτη θεωρεί ότι η οικονομία ε, και τα κέρδη των ε, απομιμήσεων φτάνουν στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ ε, που ισοδυναμεί με το ΑΕΠ 150 μικρών χωρών. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας λοιπόν, ε, συντομία. Θα, θα διασκεδάσω όσο μπορώ τις ανησυχίες σας. Ελπίζω να με βοηθήσετε με την υποστήριξή σας να υλοποιήσω το στόχο μου. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα περνάμε στις παρεμβάσεις των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Σαΐφη για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Από την έναξη ισχύω τη συνθήκη Αβωνά, ε, το Κοινοβούλιο έχει καινούριε εξουσίε που θέλουμε να την χάνουν σεβασμού ήδη από τώρα. Ακούσαμε τον Επίτροπο και του ζητάμε να ξεκινήσει μια διαδικασία μόνιμης διαβούλευσης και που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια για το θέμα της άκτα. Έτσι ώστε το Κοινοβούλιο και αυτοί τους οποίους εκπροσωπούμε να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με σεβασμό βέβαια στην ρήτρα της εμπιστευτικότητα, όπως μας είπατε. Χρειάζεται είναι και είναι ο μόνος τρόπος αυτός για να καταφέρουμε να συμμετάσχουμε και εμείς όπως πρέπει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Η ομάδα μου και εγώ ίδια σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταλήξουν σε μια πολυμερή συνθήκη που θα βελτιώνει τις προδιαγραφές εφαρμογής, που θα κάνει σεβαστά τα ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ε, και στην, την οποία επίση να προσυπογράψει και η Κίνα και άλλε ανερχόμενε οικονομίε. Η παραποίηση είναι μια μάστιγα αυτή τη στιγμή. Οδηγεί σε αθέμητο ανταγωνισμό και πλήττει την οικονομία, την κοινωνία αλλά και το πνεύμα. Διότι στερεί από τους δημιουργούς και από τις επιχειρήσεις τα δικαιώματά τους. Επιχειρήσεις και δημιουργοί που έχουν επενδύσει πολύ χρόνο και προσπάθεια και εμποδίζει τη δημιουργικότητα στο μέλλον. Ταυτόχρονα πλήττει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι με την ανάπτυξη του δικού μας ψηφιακού περιβάλλοντος δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η παραποίηση έχει γίνει άειλη. χωρίς, ε, μάλλον με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, θα πρέπει να διώξουμε αυτούς στο ίντερνετ που παραβαίνουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. David Martin. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη συνδρομή σας διότι είπατε ότι στο τέλος είχατε ανησυχίες και απαντήσατε μέχρι κάποιο σημείο, Δεν με έχετε πείσει πλοίο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις άκτα. Έχουμε κοινά σημεία, πρέπει όμως να υπάρχει κάλυψη των συμφερόντων. Η παραποίηση είναι εις βάρος και της δημοσίας υγείας. Εμείς συμφωνούμε με την επίθεση κατά της πειρα και της παραβίασης των ε, πνευματικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει όμως κανείς να έχει όρια. Όταν λοιπόν ε, μου δίνεται μία ε, πλήρη βεβαίωση το δέχομαι αλλά νομίζω ότι θα κοιτάξετε να μου ξεφύγετε από την πίσω πόρτα. Δέχομαι όμως αν μου λέτε ότι θα παραμείνει σεβαστό το πλήρω στο στο και εκτιμένο. Εδώ όμως ε, μας λέτε και πάλι τι θα γίνει με αυτούς που θα φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν θέλουμε το άκτα να ε, στραφεί εναντίον οποιοδήποτε για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ε, το θέμα ε, της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και του copyright δεν είναι μία λευκή επιταγή την οποία προσυπογράφουμε. Πρέπει να πιέσετε τους άλλους αλλά συγχρόνως να τους πείτε να πείτε στους ομολόγους σας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διαπραγμάτευση αν δεν έχετε ένα κείμενο το οποίο γνωρίζουμε για να μπορεί το Κοινοβούλιο να σας στηρίξει. Και ε, επίσης θα επανέλθω σε διάφορα από τα θέματα αυτά όσα θα, θα μιλήσουμε ε, για ε, τα δασμολογικά συστήματα. Ιντ Δέλτα, δυόμιση λεπτά. Προετοιμαζόμενη αυτή τη συζήτηση για το πώς θα προ, προστατεύσουμε τους δημιουργούς χρειάστηκε να θυμηθώ ότι πριν από δύο χρόνια εκλάπη ένα φορτηγό γεμάτο με αντίγραφα του βιβλίου της, του Χάρι Πότερ δύο μέρες πριν κυκλοφορήσουν. Ε, σήμερα πια ο, κάποιος δεν θα έκλεβε το φορτηγό, θα κατέβαζε ε, από το μέσο του ίντερνετ ε, το βιβλίο αυτό και θα το, ε, θα το κυκλοφορούσε με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονό ότι οι διαπραγματευτέ χρειάστηκε να, υπογραμμίσουν, να υπογράψουν μια ε, ρήτρα μη αποκάλυψη, είναι ψευδές. Ε, η δική σας δήλωση ήταν τελείω διαφορετική. Αν δεν υπάρχει μια τέτοιου είδου ρήτρα, τότε όλα τα ε, σχετικά έγγραφα θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Αν όμως υπάρχει μια τέτοια ρήτρα, Θέλουμε η Κομισιόν να μα πει πώ θα εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια και πληροφόρηση του κοινού, όχι μόνο του Κοινοβουλίου. Γιατί η περιορισμένη πρόσβαση, ε, ε το να δοθεί περιορισμένη πρόσβαση στο Κοινοβουλίο δεν αρκεί. Η κοινή γνώμη είναι, έχει δικαίωμα να γνωρίζει κάτι θα την επηρεάσει. Τέτοιου είδου συμφωνίε, έτσι και αλλιώ, ε, τέτοιου ρήτρε, θα πρέπει να μην επαναλαμβάνονται στο μέλλον η, η, η δημοκρατική συνομοποίηση ε, είναι πολύ αδύναμη. Δεν, ε, η διαπραγματευτική συντολή δεν έχει λάβει έγκριση από το Κοινοβούλιο. Εντάξει, θα μας πείτε, δεν προβλέπεται από τον νόμο. Εντάξει, αλλά δεν είναι ηθικό. Γιατί δεν είναι δυνατόν 27 υπουργοί να δίνουν άδεια εξουσιοδότηση στην Κομισιόν να διαπραγματευτεί εξ ονόματο όλων των πολιτών τη ευρωπαϊκή Ένωση, κανόνε του οποίους δεν γνωρίζουμε, το Κοινοβούλιο διαφωνεί με ε, ε τακτικούς ελέγχους στα λάπτοπ, ε, αβάσιμες ποινές ε, και τιμωρίες κλπ. Λοιπόν, καλό ταξίδι στην Ισλανδία τον επόμενο μήνα κύριε Επίτροπε, και φροντίστε το iPod σας να μην περιλαμβάνει ε, υλικό το οποίο έχετε καταβάσει από το Internet παράνομα. Ευχαριστώ κύριε Ινφελτ. μισή λεπτό, Έγκστρομ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν που επιτέλους κατάφερε να μιλήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά από δεκαετίες και να ενδιαφερθούν οι πολίτες για αυτό το θέμα της ΑΚΤΑ. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να επικρίνω την Κομισιόν για τη μέθοδο που χρησιμοποίησε. Ε, παρακολουθούμε τις ε, διαπραγματεύσεις και είμαστε έξαρλοι που θέλετε να περιορίσετε την ελευθερία και την επιχειρηματικότητα γιατί το ζητάνε κάποιες ε, μεγάλες εταιρείες. Ε, είμαστε έξαλλοι που δεν υπάρχει καθόλου διαφάνεια. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα έτσι σε μια δημοκρατία. Αύριο θα ψηφίσουμε ένα ψήφισμα που ζητάει από την Κομισιόν να σεβαστεί τη συνθήκη και να βάλει όλα τα έγγραφα άκτα επιτάπητο. Ελπίζω να υιοθετηθεί με συντριπτική πλειοψηφία το ψήφισμα αυτό. Το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα, το δικαίωμα στην πληροφόρηση ε, είναι θεμελιώδη στοιχεία μιας ανοιχτής ε, κοινωνία. Αύριο θα δείξουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να σεβαστεί αυτά τα δικαιώματα στην εποχή της πληροφορία. Θα θέλαμε ε, αυτή την πληροφορία, νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας. Και θα υπενθυμίσουμε στην Κομισιόν ότι εδώ είμαστε κοινοβούλιο και δεν είμαστε τίποτα ουτιδανοί που θα πρέπει να μας αγνοήσετε. Ευχαριστώ σνικ για δύο λεπτά. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον Κάρελ Ντεγκούχτ διότι ε, επέτυχε μία πρόοδο σε σχέση με τους προκατόχους του που δεν ε, έδιναν σημασία στο κοινοβούλιο και δεν το ενημέρωναν. Αλλά τώρα αμφιβάλλω διότι ελέγχθη ότι πρέπει να σεβόμαστε τις σοβαρές προσωπικότητες προηγουμένως όμως όταν μιλούσε ο κύριος Καμάλ ο ο Επίτροπος καθάριζε τα γυαλιά του. Ε, θα έπρεπε η πνευματική ιδιοκτησία να γίνεται πιο σεβαστή από ότι στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων άκτα διότι υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα και άλλες οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και ε, θα ήθελα να κάνω μία έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι εκπρόσωπος των κρατών μελών και ε, προσωπεί τα κράτη στις διαπραγματεύσεις ότι δεν πρέπει η συμφωνία αυτή να γίνει μία γκυλοτήλα και να μην καταστρέψει ε, τις, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για software στην Ευρώπη. λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, από τη μία είμαι έκπληκτη και από την άλλη ανήσυχη όταν βλέπω ότι η Κομισιόν υπερασπίζεται την εξή θέση. Ότι δηλαδή μπορούν να γίνουν έστω και μερικώς διαπραγματεύσεις μυστικές. Όταν πρόκειται για νομοθεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, για τις ε, θεμελιώδεις προσωπικές ελευθερίες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η Κομισιόν λέει ότι μπορούν να μείνουν μυστικές πληροφορίες τέτοιου τύπου που αφορούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών. Εγώ ζητώ να σταματήσουν διαπραγματεύσεις και να ξαναρχίσουν μόνο όταν οι υπόλοιποι εταίροι στις διαπραγματεύσεις είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν με πλήρη διαφάνεια. Είναι μία από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Διαφάνεια. Διαφάνεια, κύριε ε, Επίτροπε, ιδίω όταν πρόκειται για θεμελιώδεις, ε, θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα. Όλα τα χαρτιά πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι όλα τα χαρτιά πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Ευχαριστώ κυρία Σβένσον. Τώρα, Στάσεν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν ένα θέμα συζητείται και κλεισμένο το θυρών, αρχίζουν και χτυπάνε καμπανάκια. Όπως σε αυτή, σε αυτή την περίπτωση, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται. Όταν μαγειρεύονται πράγματα πίσω από κλειστέ πόρτες, μας ανησυχεί. Γιατί, γιατί οι πολίτες δεν μπορούν να πούν τη γνώμη τους. Πρέπει να μπορούν να προβλέψουν τι φαγητό θα μαγειρευτεί. Για να μπορούμε να πούμε για τη γνώμη μας. Το Κοινοβούλιο και οι πολίτε πρέπει να ενημερώνονται. Αυτό που διαγράφεται στο μέλλον για την άκτα μας ανησυχεί. Ιδιαίτερα τα όσα προβλέπονται για το ίντερνετ. Κινδυνεύουν οι ελευθερίες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Παραβιάζεται και η αρχή της επικορικότητας. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα έχουν τίποτα πλέον να πούνε για αυτό το ζήτημα. Ζητούμε διαφάνεια και διαφωνούμε με την ποινικοποίηση των πράξεων των πολιτών. Τα κράτη μάλιστα παρακολουθούν ως θεατές. Η Κομισιόν από την άλλη μεριά τι κάνει μέσα σε αυτή την κουζίνα που μαγειρεύει και γιατί οι αμερικανικές επιχειρήσεις είναι μέσα στην κουζίνα. Τι κάνουν εκεί πέρα προσπαθούν να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα φαντάζομαι, αλλά τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών είναι λιγότερο σημαντικά. Εμείς μαχόμαστε για τα συμφέροντα των πολιτών. Το κόμμα μου διαφωνεί ασφαλώ με την παραποίηση ή με τα ε, παραποιημένα φάρμακα. Δυστυχώ όμω δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επειδή δεν ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στι διαπραγματεύσει. Παραβιάζεται, παραβιάζονται τα δικαιώματά μας ως ε, ευρωβουλευτών. Όλα γίνονται πίσω από κλειστέ πόρτες. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Σουζάννα Ρόιτοβα. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Η παγκοσμιοποίηση και η προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα διότι κατακλυζόμαστε από παραποιημένα προϊόντα που είναι επικίνδυνα για την ε, υγεία των πολιτών και ε, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οι αρχές διότι ε, δεν δεν υπάρχει επαρκής μηχανισμός εποπτικός ούτε καν υψηλές κυρώσεις για τους παραποιητές ε, πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να βελτιωθεί. Δεν είναι όμως ε, ε, στόχος μας συγχρόνως να τιμωρούμε το μαθητή που κατεβάζει κάποιο στοιχείο από το ίντερνετ. Θα πρέπει να προστατευθούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων για να μπορούν να διαφυλαχθούν οι προσωπικές τους ελευθερίες και ε, θα πρέπει ε, γέρος επιπλέον Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για ε, το θέμα του SWIFT. Δεν θέλω να μας φέρνετε πρώτε τελεσμένων γεγονόταν εάν δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες ανησυχίες των πολιτών μας. Εδώ όπως ξέρετε η Κίνα είναι ένας από τους προτεργάτες των παραποιήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι μέτρα λαμβάνονται και αν διαπραγματεύεστε με την Κίνα για να προσυπογράψει αυτή τη συμφωνία. Σου στα δύο λεφτά, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες για να παραμείνει η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο ε, συνδέονται με την ε, επανακίνηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, στον παραγωγικό ιστό μας, την ικανότητα να κατακτήσουμε νέες αγορές. Όλα αυτά είναι εκ των ε, Σε αυτό το πλαίσιο η καταπολέμηση των απομιμήσεων είναι πολύ σημαντική. Η προστασία των εμπορικών σημάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι μη οικονομικά εργαλεία για να αποκτήσει το σύστημά μας ανταγωνιστικότητα. Είναι όμως και συγκεκριμένα παραδείγματα των, της αρχής της δημοκρατικότητας στον εμπορικό τομέα ε, του σεβασμού των κανόνων, κανόνες που ποδοπατήθηκαν τα τελευταία χρόνια ε, στα πλαίσια της διεθνούς ε, κερδοσκοπίας. Η άκτα είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της, καταπο, της παραποίησης που έχει φτάσει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο ε, και συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και που ε, θέτει εν αμφιβόλο τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου όπως αυτό της υγείας, αν σκεφτούμε ας πούμε τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Μην ξεχνάτε λοιπόν αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο. Ε, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε όμως και το σεβασμό κάποιων βασικών αρχών δεν μπορούμε να κρύψουμε την ανησυχία μας για τη νομική βάση της ε, συνθήκης, για τη διαπραγματευτική εντολή, για την έλλειψη διαφάνειας. Ποιος, ε, ε, εμείς εκπροσωπούμε 500, εκατομμύρια πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερωνόμαστε. οι διαπραγματευτές οι διαπραγματευτέ τη Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο για την πρόοδο των εργασιών και θα πρέπει να μας ενημερώνουν ούτω ώστε να κάνουμε πλήρη αξιολόγηση. Μόνο με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλού η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναπτύξει καλύτερα το δυναμικό της. Το ψήφισμα πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ακριβώς γι' αυτό πρέπει να υπερψηφιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σούστα. Αλεξάνδρ Άλβαρο για δυόμιση λεπτά. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Ντεμπούχτ, έχετε αναλάβει μία βαριά κληρονομιά και ε, θα πρέπει να αντεπεξέλθετε στις διαπραγματεύσεις άκτα ε, χωρίς να υπάρξουν υπεκφυγές διότι ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την υγεία των πολιτών μας και επίσης να αποφύγουμε τις τις ζημίες οι οποίες οφείλονται στην κυκλοφορία των παραποιημένων προϊόντα και ανέρχονται σε πολύ μεγάλα ποσά. Οδηγούν επιπλέον σε ζημίες και ε, σε απώλεια θέσεων, δεν είναι δηλαδή προς συμφέρον μας. Για τα φάρμακα υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των πολωτών και αυτό δεν είναι μία παραδεκτή ε, κατάσταση. Ε, Πρέπει λοιπόν να διαπραγματευτούμε, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ε, το, η εντολή διαπραγματεύσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σέβεται ε, το κοινοτικό κεκτημένο και δεν θα υπάρξει μία παράδεκτη συμφωνία που θα αποτελέσει την κατάληξη και ε, επιπλέον θα πρέπει να μας υποβληθεί και θα μας ζητηθεί η γνώμη μας. Με άλλα λόγια το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί πλήρη διαφάνεια και την δημοσίευση όλων των διαπραγματευτικών εργάφων. Ε, Εάν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να προχωρήσει πρέπει να ενημερώνει και για μένα τίθενται τρία βασικά θέματα. Αφενός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει εφαρμογή ενός συστήματος το Three Strikes διότι αυτό θα είναι αντίθετο με τις αποφάσεις μας σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δεύτερον, η Επιτροπή μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει μία συμφωνία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα είναι αντίθετη με τα συμπεφωνημένα μας. Και τρίτον, ε, πρόκειται να δεχθεί θέματα τα οποία ξεπερνούν τις αρμοδιότητές της και τα οποία δεν θα μπορούμε να ελέγχουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Άλβαρο. 1,5 λεπτό, Άλμπρεχτα. Κύριε Ντεγκούχτ, πριν από ένα χρόνο, λίγο παραπάνω χρόνο, είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊ... σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει διαφάνεια των διαπραγματεύσεων και να περνούν όλα τα θέματα από το Κοινοβούλιο και ε, να μπορέσουμε να σεβαστούμε και την ε, καταπολέμηση των παραπίσεων. Τι κάνατε από όλα αυτά, τίποτα. Μαζί με την ε, ε, συμμαχία σας διαπραγματεύεστε με κρυφή διπλωματία σε πάρα πολλούς τομείς πέραν των ισχυών των ε, κανόνων και της εντολής την οποία έχετε. Δεν μας ενημερώνετε για τίποτα αλλά πήγεται το σκάνδαλο διότι από την 1η Δεκεμβρίου δεν μπορείτε πλέον ε, να μας αγνοείται διότι οι πολίτες φρόντισαν με τη συνθήκη της Λισαβόνας επιτέλους να υπάρξει κάποιος φραγμός. Τι κάνετε λοιπόν, σαν Επιτροπή είσαστε ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Πρέπει να φροντίσετε όλα να γίνονται σεβαστά. Και αν δεν μπορείτε να το εγγυηθείτε θα πάρετε από αυτή, αυτό το κοινοβούλιο μία αρνητική απάντηση και αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε ε, ότι θα διαπραγματευτείτε κάτι προς όφελός μας τότε σταματήστε τις διαπραγματεύσεις στο θέμα του ΆΚΤΑ Ευχαριστώ Λέω Ερικ ένα λεπτό Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε Όλοι μας είμαστε αντίθετοι με την παραποίηση και τις απομιμήσεις και, αλλά μας ε, είπατε ένα παραμύθι για μικρά παιδιά, ε, κύριε Επιτροπέ, για να δικαιολογήσετε ότι διαπραγματεύεστε μια διεθνή συμφωνία πίσω από τι πλάτε των λαών και των εκπροσώπων του. Σα υπενθυμίζω, κύριε Επιτροπέ, ότι το άρθρο 218 τη συνθήκη τη Λισαβόνας αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Με τη συμφωνία ΑΚΤΑ εμπίπτουμε ακριβώ σε αυτό το άρθρο. Λοιπόν, σεβαστείτε τα λόγια σας και τη συνθήκη σας. Μόνο να ανησυχούμε μπορούμε για, το, για τις ε, θεμελιώσεις ελευθερίας. Τελικά, έτσι όπως πάτε, ε, οι επιχειρήσεις θα είναι αυτές που θα επιβάλλουν κυρώσεις. Απ' την άλλη μεριά, <laughs> οι ε, συνοριακές διατελωνιακές αρχές ε, άλλων χωρών θα μπορούν να ψάχνουν μέσα στις, ε, στις ε, βαλίτσες μας και τις αποσκευές μας ε, για να βρουν παραβάτες. Και το SWIFT υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται για την τη τρομοκρατίας και είδατε ε, πώς το ε, υπερνικήσαμε, το νικήσαμε, το ίδιο θα κάνουμε και με την άκτα. Γιατί η άκτα αυτή τη στιγμή προσβάλλει τα, ανθρώπινα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θέλουμε να δούμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κριστιανά Μουσκαρδίνη για δυόμιση λεπτά. Ε, Χριστιανά Μουσκαρδίνη. Η συμφωνία άκτα είναι σημαντική για να υπάρξει πλήρης εναρμόληση ε, των εμπορικών αμυντικών μέτρων στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία και την απομίμηση. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν ευαίσθητα θέματα όπως και είναι σημαντικό να εφαρμοστούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, να προστατευτούν τα δεδομένα. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Η Κομισιόν θα πρέπει να δεσμευτεί 100%. Θα πρέπει να σεβαστεί το επίπεδο εμπιστευτικότητας και τα διαπραγματευτικά κείμενα θα πρέπει όμως να δοθούν στη διάθεση του Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να παρακολουθεί το Κοινοβούλιο τις συμφωνίες και να κάνει παρατηρήσεις αν χρειάζεται στους συμμετέχοντες διαπραγματεύσεις άκτα. Ε, ε, κύριε Επίτροπε, αυτά που μα είπατε μας κάνουν να ελπίζουμε, αλλά θα θέλαμε μετά τα λόγια να ακολουθήσουν τα έργα. Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν ε, πολέμησε για να υπερασπιστεί του Ευρωπαίους ε, παραγωγούς και τους καταναλωτές από την απομίμηση και από μέτρα καταλέμηση και παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας στο ίντερνετ. Θα εξακολουθήσουμε λοιπόν να είμαστε ενεργοί στις διαπραγματεύσεις Δυστυχώς όμως ε, θα θέλαμε η Επιτροπή να καλέσει και άλλες χώρες πέρα από τις 12 που συμμετέχουν. Ελπίζουμε όλο και περισσότερες χώρες να εμπλακούν, αναπτυσσόμενες χώρες, αναδυόμενες χώρες, να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και να προσυπογράψουν τελική συμφωνία. Ούτως ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη, μια πιο πλατιά ε, εφαρμογή για να καταπολεμήσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την απομίμηση και την πειρατεία. Είναι μια οικονομική μάστιγα που ε, σκοτώνει πολλούς παραγωγικούς τομείς. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν σήμερα ε, να προστατεύσουμε τους καταναλωτές που εκτίθενται σε διάφορες ζημίες, μεταξύ των οποίων και προβλήματα και ζημίες εναντίον της υγείας τους. Αν δεν υπάρχουν καθαροί κανόνες, αγαπητέ Επίτροπε, και για το ίντερνετ, το ίντερνετ στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον όλων μας. Όλοι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι, ό,τι μπορούμε για να το εμποδίσουμε αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο ατομικής ιδιωτικής σφαίρας, αλλά και ασφάλειας των χωρών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μουσκαρδίνη. 1,5 λεπτό, ε, Εμινέ Μποσκιούρτα. Μια συμφωνία που έχει ε, συναυθεί και κλεισμένο το θηρόν δεν είναι αυτό το οποίο ζητούν οι πολίτες μας. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν διαπραγματεύεται μια σημαντική εμπορική συμφωνία, την άκτα και κλεισμένο των θηρών. Σε καμία χρονική στιγμή ούτε τα Εθνικά Κοινοβούλια ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν καταφέρει να ασκήσουν δημοκρατικό έλεγχο για το περιεχόμενο των συζητήσεων. Διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα μέσα στο σκοτάδι οι πολίτες για μία ακόμα φορά είναι, ε, βρίσκονται εκτός. Και εδώ δεν πρόκειται για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Συμφωνώ. Η ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει να αναθερμανθεί και η ε, πνευματική διοκτησία αποτελεί ένα κομμάτι. Αλλά ε, αυτή η μυστικοπάθεια δεν βοηθάει. Άλλωστε δεν ξέρουμε καν αν ο Επίτροπος Εμπορίου και Εμπορικών Σχέσεων συνεργάζεται με την Επίτροπο ε, που έχει στην αρμοδιότητά της τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα ληφθεί υπόψη η γνώμη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Το και τώρα Λίχτεμπεργκερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κατά τις ακροάσεις για τη νέα επιτροπή υπήρχε ε, η διαφάνεια μία από τις αρετές τις οποίες ε, απαιτήσαμε. Ε, εσείς σήμερα μας είπατε ότι όλα είναι σχεδόν διάφανα και ανοιχτά αλλά δυστυχώς εγώ δεν παρακολουθώ αυτό τον ορισμό της διαφάνειας και το ίδιο ισχύει και για ένα μεγάλο αριθμό των συναδέλφων μου ευρωβουλευτών διότι διαφάνεια είναι κάτι διαφορετικό από ε, ε, μερικά ψίχουλα ε, πληροφοριών που μας δίδονται λέγοντας ότι δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα άλλο γιατί έχουμε υποσχεθεί σε κάποιον ότι θα μείνουν μυστικές οι διαβουλεύσεις. Δεν είναι όμως δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε τυφλά προς διεθνείς συμφωνίες για να συμφωνήσουμε με εμπορικούς εταίρους οι οποίοι θα επηρεάσουν ε, το μέλλον μας. Αυτό δεν είναι πλέον ε, εφικτό μετά την ε, ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Διότι εάν υπάρχουν κρυπτά και αδιάφανα τα θέματα θα παραμείνουν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε αξιοπιστία για την προστασία της καινοτομίας στην οποία προβάλλεται. Δεν θα υπάρξει όμως αξιοπιστία αν όλα γίνονται και κλεισμένων των θυρών και μετά προσπαθείτε να καθησυχάσετε τους άλλους ότι τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο τρομερά. Δεν είναι η σωστή οδός αυτή κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Λίχτεμπέργκερ. Και τώρα, Κατρίν Τροτμάν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Α το πούμε ξεκάθαρα. Ο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσει για την εμπορική συμφωνία κατά των απομιμήσεων δεν είναι σωστό κατά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί ω νέοι συνομοθέτε σε αυτόν τον τομέα, με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, έχουμε το δικαίωμα να ενημερωνόμαστε πλήρω. Και παράλληλα με αυτή την πληροφορία που δέχεται το Συμβούλιο. Τα κείμενα που ε, λάβαμε μας απέδειξαν ότι η διάσταση αυτή δεν γίνεται σεβαστή. Τώρα επί της ουσίας. Η αγορά των απομιμήσεων ε, επίσης ε, στο ίντερνετ ε, περνάνε στο ίντερνετ επίσης υπάρχουν προβλήματα ε, υπάρχουν, υπάρχει αντιστροφή του βάρους της ευθύνης ε, υπάρχει ε, παραβίαση της ε, συμφωνίας του e-commerce αλλά και των, και των δικαιωμάτων των πολιτών. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη δείξει ότι ενδιαφέρεται για αυτές τις αρχές καταψηφίζοντας τη συμφωνία SWIFT. Μπορούμε να το ξανακάνουμε. Θέλω να τονίσω τη σημασία του ψηφίσματος που συζητάμε σήμερα και συγχαίρω τον εισηγητή μας που στέλνει ένα συμβολικό ε, μήνυμα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε ε, στο Catch the Eye. Ένα αίτημα έχουμε, ένα λεπτό, στον κύριο Γιώργο Παπαστάμκου. Παπαστάμκο. Όντων δεν πλήττει μόνο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά ενέχει και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της εφαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων εμπορικών εταίρων στη συζητούμενη πλειονομερή συμφωνία είναι ζητούμενο. Η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πρέπει να συμμορφώνεται πλήρω με το σχετικό κεκτημένο, κοινοτικό κεκτημένο, να σέβεται τι θεμελιώδει ελευθερίε και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να διασφαλίζει την ελεύθερη ροή πληροφοριών και να μην επιβαρύνει αδικαιολόγητα τι νόμιμε εμπορικέ συναλλαγέ. Τέλο, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση καθ' όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης τηρουμένης της εύλογης εμπιστευτικότητας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Παπαστάμκο. Φερέιρα, ένα λεπτό. Η διαδικασία είναι πολύ σκοτεινή Υπάρχει όμως κάτι το οποίο αναφαίνεται. Προσπαθούμε να διευρύνουμε τα δικαιώματα πνευματικής διοξίας των επιχειρήσεων για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αγνοώντας δημοκρατικούς κανόνες, αγνοώντας τον κανόνα της διαφάνειας, εκτός οποιοδήποτε δημοκρατικού ελέγχου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αν χρειαστεί, περιορίζεται ακόμα και η συνολική πρόσβαση σε αγαθά πρώτης ανάγκη όπως φάρμακα. Επίσης παραβιάζεται τα δικαιώματα ε, ιδιωτικής, ε, της ιδιωτικής ε, σφαίρας ή της πρόσβασης σε πληροφορίες. Η της προσβασης σε η προασπιση των οικονομικών συμφερόντων επιχειρήσεων και τομέων δεν συμβιβάζεται με την προάσπιση των δημόσιων αγαθών. Τα αποτέλεσματα αυτή της πολιτικής είναι καταφανή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φερέιρα. Και κλείνουμε με τον Επίτροπο Ντεχούχτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας τις παρεμβάσεις μετά από την πρώτη μου παρέμβαση σκέφτηκα ότι πολλοί από εσά δεν ακούσατε αυτά που είπα. Γιατί ξεκαθάρισα στην πρώτη μου παρέμβαση ότι θα σεβαστούμε το κοινοτικό κεκτημένο. Είπα ήδη ότι θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω ότι οι άλλοι εταίροι που συμμετέχουν ε, στην, ε, στις διαπραγματεύσεις δίνουν το πράσινο φως για την ε, δημοσιοποίηση των κειμένων επί των οποίων διαπραγματευόμαστε. Και ξεκαθάρισα ότι αυτό θα αφορά μόνο τις εμπορικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα μπορούσα να πω κι άλλα για αυτά που δεν ακούσατε. Επομένως, δεν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που μου απευθύνατε. Γιατί νομίζω ότι στην πρώτη μου παρέμβαση σας έχω ήδη καλύψει. Ο David Μάρτιν ρώτησε τι γίνεται αν κάποιος όχι φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από, τη χώρα, από μια χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνία Άκτα. Ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί φυσικά εξαρτάται αυτό που πηγαίνει. Αν πηγαίνει σε μια χώρα όπου δεν έχει προσυπογράψει την Συμφωνία Άκτα, εξαρτάται από την αστυνομία και τα τελωνία της εν λόγω χώρα. Και αυτό είναι πέρα από την ε, εξουσιοδότησή μας και την ε, αρμοδιότητά μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να προδικάσουμε θα κάνουν οι άλλοι. Δεν μπορώ να, να απαντήσω σε όλα όσα είπε η Σοφία Ιντβελτ για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Να σας πω όμως τι συμβαίνει κατά τη γνώμη μου με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το Συμβούλιο δίνει μια διαπραγματική εντολή στην Κομισιόν, η Κομισιόν διαπραγματεύεται και το Συμβούλιο λαμβάνει μια απόφαση για την εντολή αυτή με βάση τους δικούς του εσωτερικούς κανόνες. Και αν ένας υπουργό, το Συμβούλιο Υπουργών, χρειάζεται την έγκριση από το Εθνικό του Κοινοβούλιο, αυτό δεν είναι θέμα ευρωπαϊκού δικαίου. Το, αυτό το προβλέπει το εθνικό δίκαιο, η εθνική νομοθεσία. Και όλα αυτά τα πράγματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στη χώρα σας, ας πούμε, για πολλά τέτοια θέματα χρειαζόσαστε ούτως ή άλλως την ε, σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν πρέπει να κρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει το Συμβούλιο. Μια, αν το Συμβούλιο σέβεται τη ε, συνθήκη και τους εσωτερικούς του κανονισμούς, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν καλώς. Ε, με προστατεύετε, λέτε ότι δεν θα πρέπει να ελέγχει κανένα το iPod μου. Σας ε, διαβεβαιώ, δεν έχω ακόμα αγοράσει iPod. Και δεν θα πάω και στη Νέα Ζηλανδία. Αφήνω τους υπαλλήλους. Έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο. Τώρα, τη συζήτηση για την κουζίνα την αφήνω στην κυρία Στάσεν. Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα στο οποίο θα απαντήσω αφορά την Κίνα. Κυρία Ρόιτοβα, η Κίνα δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, η Κίνα είναι η πρώτη διδάξα διδάξασα στις απομιμήσεις. Έχουμε πάρα πολλές διαπραγματεύσεις και συζητήσεις εν εξέλιξη με την Κίνα, ειδικά στα πλαίσια του οικονομικού διαλόγου και έχουμε πολλές ε, φορές τονίσει τα θέματα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για το εμπόριο μέσω ίντερνετ αλλά και στα πλαίσια άλλων αρμοδιοτήτων, ε, δραστηριοτήτων. Η άκτα όταν ολοκληρωθεί θα είναι ανοιχτή για να προσυπογραφεί από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Και ελπίζω να την προσυπογράψει για το καλό της βιομηχανίας της και η Κίνα. Θα ήταν καλύτερο και η Κίνα να έχει μια καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κοιτάξτε τι γίνεται με άλλες χώρες, όπου στο παρελθόν ε, έκαναν ακριβώς το ίδιο. Σήμερα υπάρχει μια καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν συμφωνώ με την κυρία Ιαρή και με την κυρία Τρότμαντ για το άρθρο 218. Αυτό το άρθρο λέει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Μα ενημερώνεστε αγαπητοί βουλευτές και με το παραπάνω. Αυτό που κάνουμε για την ενημέρωση ξεπερνάει κατά πολύ τα όσα λέει το άρθρο 218. Κατά πολύ. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Το είπα και στην αρχική μου παρέμβαση. Θα επιμείνουμε, ότι, θα επιμείνουμε να δώσουν το πράσινο φως και όλες οι υπόλοιπες χώρες, ούτω ώστε να δημοσιοποιήσουμε το σημερινό σχέδιο κειμένου. Και δεν είναι σωστό να λέτε ότι δεν σεβόμαστε το άρθρο 218. Και λέω εν παρόδο, απευθυνόμενος προς τη Σόφη Ιντβέλτα, ότι σας στείλαμε το παράρτημα 16 που αφορά τις δηλώσεις όλων των συμβαλόμενων μερών για το σεβασμό της αρχής της εμπιστευτικότητας των εγγράφων. Ο κύριος Ντέβιτο Σάλιβαν τον Ιανουάριο του 2009 σας έστειλε τα κείμενα. Ήταν η προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, αλλά τα ίδια άτομα συναντώνται πάλι. Ο κύριος Σοσάλβα ήταν στη θέση του, κυρία Ιντβελτή ήσασταν και εσεί τότε το 2009 βουλευτή. Επομένως μην μου επιτίθεστε. Τέλος, θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι αυτό που είπα στην ακρόασή μου πρέπει να το πάρετε στα σοβαρά. Ότι θα κάνω δηλαδή ό,τι μπορώ ούτω ώστε να πάρω το ok από τα συμβαλώμενα μέρη για να συνημερώσω πλήρω. Αλλά όσο δεν έχω αυτό το ok, δεν μπορώ να σας ενημερώσω. Δεν μπορώ να σας κοινοποιήσω τα σχέδια συμφωνίας, γιατί αυτό θα παραβίαζε την εμπιστευτικότητα που υπάρχει μεταξύ μας. Παραβιάζοντας αυτή τη συμφωνία θα υπήρχαν επιπτώσεις όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις, άκτα, αλλά θα αφορούσαν και άλλες διαπραγματεύσεις με τις εν λόγω χώρες. Θα έπλητε την ίδια την εμπιστευτικότητα και θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατε και όλες τις άλλε διαπραγματεύσεις. Θα κάνω όμω ό,τι μπορώ για να σας ενημερώνω. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ανακοινώνω ότι πέντε σχέδια ψηφίσματος, πέντε προτάσεις ψηφίσματος έχουν παρουσιαστεί και με αυτό κλείνουμε αυτή τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Πάμε στο επόμενο σημείο. Και τώρα, έχουμε πάλι μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για τον κανονισμό για την εφαρμογή του συστήματος γενικευμένων τασμολογικών ε, προτιμήσεων.